κείμενο το συνοπτικό πρακτικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ζήσαμε όλοι τα δραματικά γεγονότα ε, του Σαββατοκύριακου στην πλατεία Ανεξαρτησία ε, στο Κίεβο και είδαμε πω η Ουκρανία έζησε την πιο σημαντική αλλαγή τη πρόσφατη ιστορία τη. Εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να απευθυνθώ και να εκφράσω την αλληλεγγύη μα στον ε, Ουκρανικό λαό. Θαυμάζουμε την αξιοπρέπειά τη, το κουράγιο τη και την ανθεκτικότητά τη. Γίνεται ένα αγώνα για περισσότερη δημοκρατία και δικαιοσύνη και πλήθο ανθρώπων έχασαν τι ζωέ του τι τελευταίε ημέρε. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να απευθύνω στις οικογένειες των θυμάτων τα συλληπιτήριά μας καθώς επίσης και την αλληλεγγύη μας να τους διαβιβάσω. Το Σάββατο μας ήρθε μια καλή είδηση όμως. Μετά από δυόμιση χρόνια κράτησης, επιτέλους αφέθηκε ελεύθερη η κυρία Γιούλια Τιμοσέγκο. Και σε σχέση με αυτό θα ήθελα Ρίτα, να ευχαριστήσω τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατ Κόξ, και τον πρώην πρόεδρο της Πολωνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Αλεξάνδρε Κβασιεύσκη, και να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Ε, έπαιξαν ένα ρόλο πρωταγωνιστικό για να αφαιθεί ελεύθερη η κυρία ε, Τιμοσέγκο. Η Ουκρανία, κυρίε και κύριοι, είναι ενώπιον τεράστιων προκλήσεων. Ήψιστο στόχο θα πρέπει να είναι η σταθερότητα και η ενότητα τη χώρα, καθώ επίση και αποκατάσταση τη εθνική συμφιλίωση. Γι' αυτό θα πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που να συνενώνει ε, τις διάφορες δυνάμεις της χώρας και να προετοιμάσει τις ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές της 25ης Μαΐου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνή κοινότητα οφείλουν να είναι στο πλευρό του λαού για να αποτραπεί η επαπειλούμενη οικονομική κατάρρευση της χώρας και να επανέλθει ε, η Ουκρανία σε μια σταθερή δημοκρατία. Σήμερα το βράδυ επιστρέφει ad hoc αντιπροσωπείο μας από το Κίεβο και θα φέρει τις νέες εντυπώσεις. Την Τετάρτη θα ασχοληθούμε στην Ολομέλεια εκτενώς με το θέμα αυτό. Κυρίες και κύριοι, σε αλληλεγγύη με τους ανθρώπους εκεί αλλά και σεβόμενοι τα θύματα που έπεσαν στον αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία και άφησαν και τη ζωή τους, σας παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Κυρίες και κύριοι, πριν από δύο έτη και πλέον, στην Κεράλα έγινε τραγικό ναυάγιο. Δύο Ινδοί ε, έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, ο Μασιμιλιάνο Λατόρε και ο Σαλβατόρε Τζιρόνε, Ιταλοί, ε, ναυτικοί ε, βρίσκονται στα χέρια της συνδικής Δικαιοσύνης. Ε, δεν θέλω να πω στην ουσία του θέματος, εάν ευσταθεί η κατηγορία, αλλά θέλω να εκφράσω τις ε, δικές μας ανησυχίες και να συμφωνήσω με την Ιταλική κυβέρνηση. Καλώ τις συνδικές Αρχές εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αμελητή να εφαρμόσουν το δικαίω, ε, της και το διεθνές δίκαιο. Η καταπολέμηση της πειρατείας είναι ε, κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε ιδιαίτερα σε απειλούμενες περιοχές. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας θα πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό ε, του κράτους δικαίου. Μόνο βάσει της διπλωματίας ε, μπορούμε και του διαλόγου να συνεργαζόμαστε. Οποιαδήποτε μορφή αντιπίνων, ε, ιδιαίτερα ε, του προκειμένου εναντίον των δύο Ιταλών πολιτών, είναι κάτι το οποίο δεν νοείται και εμείς είμαστε στο πλευρό τους και εκφράζουμε την του. Έρχομαι στις ανακοινώσεις. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στις 10 Φεβρουαρίου έγκρισε, ενέκρισε γνώμη, την εντολή